Λοιπόν, αρχίζουμε με τις εργασίες μας της Επιτροπής Ανάπτυξης. Σήμερα θα ψηφίσουμε τις τροπολογίες για τον DCI, για τον ΜΑΣ. Αλλά πριν από αυτό υπάρχει ένα άλλο σημείο στην ημερήσια διάταξη που είναι η συνεισφορά της Επιτροπής Ανάπτυξης στο σχέδιο ψηφίσματος σε σχέση με τη διάσκεψη της ΔΟΧ για την αλλαγή του κλίματος. Η Επιτροπή Ανάπτυξης έχει, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, με συγχωρείτε, έχει προετοιμάσει αυτή την έκθεση. Άρα θα πρέπει να συνταχθεί ένα βασικό έγγραφο για να αρχίσει η συζήτηση που στη συνέχεια μπορεί να αλλάξει υποτύπο τροπολογιών. Η προθεσμία υποβολής είναι 24 Σεπτεμβρίου. Επειδή το βασικό έγγραφο έχει συνταχθεί στα αγγλικά και είναι πολύ κοντά η προθεσμία, θα ήθελα να υποβάλλετε μόνο στα αγγλικά τις τροπολογίες σας. Για να βοηθήσουμε με την ψηφοφορία τη στην Επιτροπή μας που προβλέπεται για τις 10 Οκτωβρίου. Σας δίνω το λόγο για ενδεχόμενες συνεισφορές και στη συνέχεια θα ε, κάνω και εγώ ορισμένες παρατηρήσεις με τη σειρά μου. Comment s'appelle ο κύριος Πρέντα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να χαιρετήσω αυτή την πρωτοβουλία μετά από τις συζητήσεις για τη διάσκεψη της Ντόχα και θα ήθελα να συνεισφέρω και εγώ μέσα στα πλαίσια του ψηφίσματος της Επιτροπής μας και του ψηφίσματος της Επιτροπής ΕΜΒΗ. Θα αναφερθώ καταρχήν στα σημεία που φύγονται από το κείμενο και ιδιαίτερα την ανησυχία μας σε σχέση με την χρηματοδότηση των κλιματικών αλλαγών που θα περάσουν από τον προπολογισμό ανάπτυξης, περιβάλλοντος και ανάπτυξης. Συμφωνώ με το κείμενο ψηφίσματος. Θα πρέπει να βρούμε λύσεις για να αποφύγουμε τη μείωση αυτών των, αυτής της χρηματοδότησης στις υποανάπτυξη χώρες. Στη συνέχεια θα ήθελα να σας μιλήσω για το σημείο Β και Γ του προημίου διότι εδώ το κείμενο ε, στο Β λέει ότι δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε στα 100 δις που έχουν συμφωνηθεί στο Ντέρμπαν χωρίς έναν καινοτόμο μηχανισμό. Και θα ήθελα να σας υποβάλω το ερώτημα σε τι συνίσταται αυτός ο καινοτόμος μηχανισμός. Ποια είναι η φύση αυτού του μηχανισμού καινοτομίας. Θα βασιστούμε σε ιδιωτικά κεφάλαια, στον ιδιωτικό τομέα. Προβλέπουμε κάτι το συγκεκριμένο επί του θέματος. Στη συνέχεια, στο γάμα γίνεται λόγος για την ανάγκη να έχουμε πιο ε, σεβαστές ε, πηγές και αξιόπιστες πηγές για να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές. Εσείς είπατε, μιλάτε για μια νέα φορολόγηση, μια νέα μορφή φορολόγησης. Πώς μπορούμε να βρούμε τους κατάλληλους πόρους. Αυτά εν ολίγης και αναμένω τη συζήτηση γύρω από την συνεισφορά της δικής μας Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπάρτ. Στάς Μπάρτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η πρόταση αυτή μου φαίνεται αρκετά καλή. Όπως παρουσιάστηκε. Και νομίζω ότι θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε ορισμένα στοιχεία, να τα επεξεργαστούμε καλύτερα. Στο Β εμείς θα ε, ανέβρουμε, θα εξεύρουμε καινοτόμου μηχανισμούς και νομίζω ότι θα πρέπει να ενσωματώσουμε και, τον, και το τέλος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να το χρησιμοποιήσουμε σχετικά στο ε. Μιλάμε για τις δαπάνες προσαρμογής που σχετίζονται με μια γενικότερο, ένα γενικότερο έλεγχο των κλιματικών αλλαγών. Αυτό θα πρέπει να το συνδέσουμε με θέματα βιοποικιλίας, βιοπικιλότητας. Θα πρέπει να ενισχύσουμε το ε. Στο δεύτερο, στη δεύτερη παράγραφο μιλάμε για το πράσινο ταμείο, για το κλίμα το οποίο δεν πρικοδοτείται παρκώς, δεν έχει επαρκή χρηματοδότηση, γι' αυτό θα πρέπει να την ενισχύσουμε. Στο σημείο 3, εμείς, εμάς μας απασχολεί, είμαστε πράσινοι, αλλά και ως Επιτροπή Ανάπτυξης θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να προωθήσουμε και να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των αυτοχθόνων και η αποψήλωση των δασών θα πρέπει να σταματήσει. Και αυτό θα τα προωθήσουμε μέσω τροπολογιών. Κύριε Γκέρνς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να σας υπενθυμίσω καταρχήν ότι παίζουμε ένα μάλλον περιθωριακό ρόλο εδώ, γιατί το θέμα αφορά κυρίως την κλιματική αλλαγή και το πώς επηρεάζει τις ε, αναπτυσσόμενες ε, χώρες ε, είναι αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς. Νομίζω ότι ο κ. Πρέντα έθεσε τον δάκτυλο στον τύπο των ύλων. Χρειάζεται πραγματικά καινοτόμα χρηματοδότηση Παρ' όλα αυτά αυτό γίνεται λίγο στερεότυπο πλέον. Το σύνδρομο του Παυλόφ ε, δεν ταυτίζεται πάντοτε με την ευφύεια. Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν κάτι διαφορετικό να λέμε. Τι μπορούμε να κάνουμε. Είπαμε, ιδιωτική χρηματοδότηση. Πολύ ωραία. Ας την συνδέσουμε με την αρχή ορυπαίνων πληρώνει. Και να δούμε ποιο είναι υπεύθυνο γιατί εδώ και στις αναπτυσσόμενε χώρε. Να εντοπίσουμε λοιπόν ε, τον υπεύθυνο της κλιματικής αλλαγή. Ε, αν θέλετε θα σα εμπιστευτώ για να συντάξετε εσεί μια τροπολογία, αλλιώ να το κάνουμε και μαζί. Και δεύτερον, κάτι που μας ενοχλεί όλους, η ανικανότητα της Ευρώπης να υλοποιήσει τις υποσχέσεις της. Γιατί τι έγινε το ε, είχαμε υποσχεθεί ένα συγκεκριμένο επίπεδο, ε, ποσοστό για την ε, αντισιακή βοήθεια και κανένας δεν το λέει πια, δεν το αναφέρει πια. Ορισμένες χώρες έχουν υπαναχωρήσει σε ό,τι αφορά την αντισιακή βοήθεια που δίδουν. Αυτό θα έχει συνέπειες σε ψηλό, σε ψηλό πολιτικό επίπεδο και κινδυνεύουμε να βρεθούμε σε μια φάση ανά ε, διανομής της βοήθειας. Δηλαδή, θα πρέπει να αποφύγουμε τα χρήματα που είχαν προβλεφθεί ε, για αναπτυξιακή βοήθεια προς συγκεκριμένε ε, χώρες ε, να ε, ξανατεθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να αλλάξει η ονομασία τους, να αλλάξει ο στόχος τους και να γίνει ο στόχος της καταπολέμησης κλιματικής αλλαγής. Ε, θα πρέπει να επιμείνουμε, να το αποφύγουμε, παρόλο ότι και η κλιματική αλλαγή είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να καταπολεμηθεί. Λοιπόν, ε, εμπιστεύομαι τον κύριο Πρέντα ε, να διατυπώσει αυτό στην τροπολογία, αλλιώ να το βοηθήσω. Ωραία, παίρνω το λόγο κι εγώ η ίδια. Θέλω να υπογραμμίσω δύο πράγματα. Σε όλα μας τα αναπτυξιακά σχέδια θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Είναι αυτό που ονομάζουμε mainstreaming του περιβάλλοντος, όπως ακριβώς κάνουμε και με το φύλλο. Όλα τα σχέδια θα πρέπει να έχουν μια περιβαλλοντική πτυχή, μια περιβαλλοντική διάσταση. Μετά να σας υπενθυμίσω ότι το 20% των εκπομπών αερίων του Θερμοκυπρίου προέρχονται από αποδάσωση, από αποψήλωση δαφθοσών και από αλλαγή χρήσης ε, δασικών εκτάσεων. Γι' αυτό το λόγο το 10% ε, ε, της ε, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στι ε, στις μεταφορές θα πρέπει να αρθεί, να καταργηθεί διότι οδηγεί σε περαιτέρω αποψήλωση γεών. Θα πρέπει επίσης να προωθήσουμε την βιολογική γεωργία και ιδιαιτέρως στις χώρες πολύ χαμηλού εισοδήματος γιατί αυτή η γεωργία, η βιολογική γεωργία συνεισφέρει στο να προλαμβάνονται οι κλιματικές αλλαγές και επίσης βέβαια βοηθάει και τους γεωργούς να βγουν από τη φτώχεια. Αυτές οι ανησυχίες πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν στο κείμενο. Ο λόγος στην Κομισιόν. Thanks. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την ευκαιρία της ανταλλαγής απόψεων με εσάς σήμερα σε αυτό το σχέδιο ψηφίσματος. Η Κομισιόν θα έλεγα ότι κατά πολύ συμμερίζεται τις απόψεις σας. Στα σημεία τα οποία μόλις αναφέρθηκαν, πιστεύω πως είναι ξεκάθαρο ότι η χρηματοδότηση θα είναι σημαντικό συστατικό στοιχείο της συμφωνίας την οποία θέλουμε να επιτύχουμε στο τέλος της χρονιάς στην Τόχα, όπως και τα προηγούμενα έτη εξάλλου από την Κοπενχάγη και έπειτα, μετά στο Κανκούν και στο Ντέρμπαν πέρυσι. Προφανώς ε, αυτό που χρειάζεται να συμφωνήσουμε για την τόχα είναι η εφαρμογή της ε, δέσμης ε, που συμφωνήθηκε πέρυσι στον Τέρμπαν και θα έλεγα πως όλα τα στοιχεία του πακέτου αυτού πρέπει να, μην, πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι δεν, να μην εστιάζουν τόσο πολύ στην ΚΑΠ. Τώρα, Εκτός από αυτή την δέσμη μέτρων θα συζητήσουμε και για την κλιματική χρηματοδότηση. Γνωρίζετε υπάρχει ένας σχετικός φάκελος ε, στο τέλος ε, φέτος του 2012 και τότε θα είμαστε στην θέση να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας όσον αφορά τη χρηματοδότηση μέχρι το τέλος της χρονιάς αλλά ταυτόχρονα να δώσουμε και ένα θετικό μήνυμα για το μέλλον. Και Τούτων λεχθέντων συμφωνώ με τις ε, παρεμβάσεις σας ε, όπου αναφέρθηκε η ανάγκη να εργαστούμε περισσότερο για την πηγή της χρηματοδότησης και να υπενθυμίσω ότι αυτό το ποσό που υποσχεθήκαμε στην Κοπενχάγη, αυτό το 1,3 ε, δισεκατομμύρια, συμπεριλαμβάνει και ιδιωτικά και δημόσια κονδύλια και οι δύο πλευρές λοιπόν καλύπτονται σε αυτήν την σε αυτό το ποσό. Φυσικά υπάρχει ανάγκη να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για καινοτομία στι ε, πηγέ μας και εμείς ως Επιτροπή συνεχίζουμε να ψάχνουμε τις επιλογές που έχουμε για διεθνεί μεταφορές ή τι μπορούμε να κάνουμε στον τομέα των αερομεταφορών, για παράδειγμα, να δούμε τι, έχουμε, ε, τι δυνατότητες έχουμε τώρα, τι εισοδήματα ή και ε, τι μπορούμε να κάνουμε στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές. Όλα αυτά θα γίνονται στα πλαίσια του G20 και εμείς χρειάζεται να συνεισφέρουμε στη διαδικασία αυτή, φυσικά. Επίσης, να συμφωνήσω και με εσάς, κυρία Πρόεδρε, για την ανάγκη να προσπαθήσουμε περισσότερο για το λεγόμενο mainstreaming και να εντάξουμε το κλίμα στην ε, ατζέντα συνεργασίας για το κλίμα. Φυσικά υπάρχει ανάγκη για περισσότερη συνεργασία με τις, ε, με τις χώρες εταίρους μας για σχεδια... δράσεις και σχεδιασμό και πιστεύω πως χρειάζεται μεγαλύτερη ανταπόκριση από μέρους μας. Και εμείς ως Επιτροπή εργαζόμαστε πολύ πάνω γι' αυτό. Κάτι τελευταίο τώρα όσον αφορά την διπλωματία για το κλίμα. Σωστά το θίξατε αυτό το θέμα στο ψήφισμα. Ξέρετε ότι ένας από τους λόγους που ήμασταν επιτυχείς στον Τέρμπαν είναι το γεγονός ότι καταφέραμε ε, να δημιουργήσουμε μια στρατηγική συμμαχία με τις ε, λιγότερο ανεπτυγμένες και περισσότερο ευάλωτες χώρες. Πιστεύω πως εξίσου σημαντικό αυτό θα είναι στην ε, επιτυχία της Ντόχα και πρέπει να προωθήσουμε αυτή την συμμαχία και να έρθουμε πιο κοντά με αυτές τις χώρες, έτσι ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα όσον αφορά την ε, ατζέντα της Ντόχα για τον πλανήτη. Μπορούμε να εργαστούμε διμερώς, περιφερειακά με αυτές τις χώρες και ε, αναμένουμε με χαρά τη συμμετοχή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας υπενθυμίζω ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι 24 Σεπτεμβρίου, ψηφοφορία στις 10 Οκτωβρίου. Θα περάσουμε στο φιλέτο της σημερινής συνεδρίασης. Ε, ψηφοφορίες σημείο 14 θα ψηφίσουμε μόνο τις τροπολογίες του χρηματοδοτικού μέσου για την αναπτυξιακή συνεργασία, προκειμένου να καθορίσουμε την εντολή μας για την διοργανική διαπραγμάτευση. Πριν περάσουμε στις ψηφοφορίες, ε, ο συντονιστή προτείνει του εξή για την διαπραγματευτική ομάδα. Μπέρμαν, εμένα την ίδια ω πρόεδρο. Monsieur Monsieur Monsieur αυτή η σύνθεση σας βρίσκει σύμφωνους για την διαπραγματευτική μας ομάδα. Ωραία, το σημειώνουμε. Σας ευχαριστώ. Η διαπραγματευτική ομάδα θα μας ενημερώνει τακτικά, κάτι που θα μας επιτρέπει να αλλάξουμε αν χρειαστεί την εντολή κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης. Αυτό θα μπορούσε να καταστεί απαραίτητο ε, κατά τη διάρκεια της ε, διαπραγμάτευσης. Ε, ας ελέγξουμε λίγο τις ε, καρτέλες της ε, ψηφοφορίας μας, τις κάρτες ψηφοφορίας μας. Κύριε Μπέρμαν, θέλει το λόγο. Ναι, πριν ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους οι συγητέ και την Κομισιόν και το Συμβούλιο για την συνεργασία τους παραδειγματική ως τώρα και το επικοδομητικό του πνεύμα. Επίση, τον Μπράιον Όχα και την Μαρή Καλέρ καθώς επίσης και την βοηθό μου. Όλοι δούλευσαν εξαιρετικά πάρα πολύ. 60 σελίδες τροπολογίες ε, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο γιατί χρειάζεται να ε, ταξινομηθούν και να δημιουργήσουν ένα αρμονικό σύνολο. Τους συγχαίρω. Euh, Προτείνω ένα τεστ, ε, μια δοκιμή των ε, καρτών. Ας αρχίσουμε τη ψηφοφορία δοκιμαστικά. Λείπει κάποιος. Μία ψήφος. Λείπει μία ψήφος. Κάποιος δεν ψήφισε. Ψηφίσατε όλοι. Ωραία. Τέλεια. Κλείνει η ψηφοφορία. Ωραία. Δουλεύει. Ξεκινάμε με την τροπολογία 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία ΦΑΜ 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 259. Όχι, συγγνώμη. Ναι, 259. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Το ελέγχουμε. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λήξη ψηφοφορία Εγκρίνεται. ΦΑΜ 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 260. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 261. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε παρακάτω. Ε, συμβασμός 9 υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 262 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 265. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 264 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται λήξη ψηφοφορίας απορρίπτεται για μία ψήφο 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Φαμ 19 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Φαμ 20 υπέρ. Κατά εποχές απορρίπτεται 266 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται τροπολογία 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 200 Είναι τα 13 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. ...268 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 32. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Φάμ 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αφέτ 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Φάμ 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 271 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Budget 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 269 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 270 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Μπάτζετ 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 272 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 273 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 274 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, budget 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται budget 20 υπέρ κατά αποχές Α, θα το ελέγξουμε ηλεκτρονική ψήφωση. Α, άρχεται Il manque Λείπει μία ψήφος. Ωραία, κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 277. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε και πάλι. Ένα της ψηφοφορίας. Λήξη ψηφοφορίας απορρίπτεται με διαφορά τεσσάρων ψήφων Σαράντα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία Τροπολογία τα δεκατέσσερα. όχι η 40 Πίπτη αν η 277 υιοθετηθεί, ε, δεν υιοθετήθηκε, ψηφίζουμε τη 40, υπέρ, 40, 40 υπέρ, κατά, ε, υπέρ, συγγνώμη, υπέρ, του εισηγητή είναι, κατά, αποχέ εγκρίνεται. Είναι τα δε... όχι, καταπίπτει, 41. 41. Υπέρ. Κατά. Αποχής. Εγκρίνεται. Είναι τα 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 280. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 281. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Κύριε Στάση, έχει το λόγο. Ehm, ε, θα ήθελα να πω ότι έχει κυκλοφορήσει ένα έγγραφο σε σχέση με τον συμβασμό 10 που θα ψηφίσουμε. Ε, είναι από τον κύριο Κάσμαν, τον κύριο Νιούτον και τον Συγητή. Θα ήθελα να προσθέσουμε κάποιες λέξεις. Αν έχετε το έγγραφο θα δείτε ποια ήταν η αρχική πρώτα συμβασμού και μετά θέλουμε να προσθέσουμε και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και με ε, ασθένειες που ε, ε, αποτελούν κίνδυνο για τη ζωή τους. Αυτά θα ήθελα να προσθέσουμε. υποβάλλουμε την, τον Πληροφορικό συμβασμό σε ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Καταπίπτει η συμβαστική πρόταση 10. Περνάμε τροπολογία ΦΑΜ 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεν θα έπρεπε να ψηφίσουμε δύο διαφορετικά τμήματα στο, στη συμβαστική πρόταση 10. Πρώτο τμήμα, δεύτερο τμήμα. δεχτήκαμε την προφορική πρόταση συμβασμού. Τώρα δεν θα πρέπει να ψηφίσουμε αν θα μπει το decent work ή δεν θα μπει. Η χωριστή ψηφοφορία θα πρέπει να έχει ζητηθεί. Μα έχει ζητηθεί. Έχει ζητηθεί. Αν πλειοψηφία θέλει να κάνουμε χωριστή ψηφοφορία, κανένα πρόβλημα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα λοιπόν. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε 24, την ψηφίσαμε. Τροπολογία 284 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία... Budget 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 287. 287. Όχι. Αφέτ 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 287 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 45 Υπέρ. Όχι. Η 44 έχει υιοθετηθεί, άρα καταπίπτει 45. Τροπολογία 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 276. Υπέρ. Όχι. Πάμε πίσω. Αφετ 18. Αφετ 18. Το πρώτο τμήμα έχει καταπέσει γιατί εγκρίναμε τη 46. Το δεύτερο τμήμα όμως πρέπει να ψηφιστεί. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας ΑΦΕΤ 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας το εξακριβώσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη ψηφοφορίας απορρίπτεται με διαφορά δύο ψήφων. 276. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Φάμ 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία, ε, συγγνώμη, συμβαστική πρόταση 11, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Είναι τα 18. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Budget 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία. Άφετ 22. Χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 295. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Budget 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Budget 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 296. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αφετ 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική εξακρίβωση. Έναξη πληροφορίας. Λείπουν λοιπόν, τρεις, δύο, δύο ψήφοι λείπουν. Λοιπόν. Μία. Λήξη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Γιατί χάσαμε τον χρόνο μας να περιμένουμε όλε ψήφους. Τροπολογία 300. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 301. Υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. Ελέγχουμε 301 εξακρίβωση, ηλεκτρονική εξακρίβωση. Άρχεται. Λήξη. Έγκρινεται. Έχω αρχίσει να κουράζομαι, είχατε δίκιο. Αφέτη 24, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Είναι τα 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 302 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ίντα... Τροπολογία budget, δεν ξέρω όμως ποιο νούμερο είναι. 25. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Είναι τα 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Budget 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 303 υπέρ κατά αποχές Α, ηλεκτρονική εξακρίβωση άρχεται λίγη εγκρίνεται με διαφορά τεσσάρων ψήφων. ΦΑΜ 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πάμε 27 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 53 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι τα 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Α, εξακρίβωση. Είναι τα 21. Σε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Είναι τα 22. Υπέρ. Κατά. ΕΠΟΧΕΣ Εγκρίνεται. Τροπολογία 306. Καταπίπτει. Ωραία. Αφέτ 25. Χωριστή σουφοριά. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Α, καταπίπτει εντάξει. Πενήντα πέντε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι τα 23. Α, είναι παρόμοιες, εντάξει. Προϋπολογισμός 27. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Προϋπολογισμός 28. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. ΦΑΜ 29. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται προπολογισμό 29 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 56 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Είναι τα 24 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Είναι τα 25 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 310 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 311 την ψηφίζουμε, λέει πρόεδρος. Il faut voter. Il faut voter. Il faut voter tous. D'accord. 311. 311 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε. 311 ελέγχουμε. Αρχίζει η ηλεκτρονική. Le vote électronique est clos. Πέρας ηλεκτρονικού ελέγχου. Απορρίπτεται με τέσσερις ψήφους διαφορά. 59 αρχίζει, μάλλον ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβασμός 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άφετ 26 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. c'était adopté et c'était adopté donc ça tombe. Amendement 61 qui est pour. 61. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προϋπολογισμός 30. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 62. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 63. Υπέρ,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 316 πέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. au 17 donc, tombe donc euh, d'accord 318 318 hyper kata αποχές απορρίπτεται. Είναι τα 26 υπέρ κατά αποχές πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά σας παρακαλώ δεν σαφές το αποτέλεσμα άρχεται η ψηφοφορία Δύο ψήφοι λείπουν. Πέρας. Εγκρίνεται. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 319 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 73 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Προϋπολογισμός 32 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Άφετ 27 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Φαμ 31 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 320 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 321 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 322 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 323 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 324 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άφετη 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται φαμ 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ΦΑΜ 34 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 328 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προϋπολογισμή 36 υπέρ, όχι, λέει πρόεδρος, έκανα λάθος. 329, 329 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 36 προϋπολογισμό περ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 330 έχει αποσύρθει της κυρία Ζαμπόρσκα. 37 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 327 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Φαμ 32. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 333 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 331 τριάντα ένα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Φαμ 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ογδόντα έξι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 Κατά πίπτη Et femmes 36. Donc, INTA 28. Καταπίπτει ίντα 28, άρα ΦΑΜ 36 ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ίντα 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Φαμ 37. Φαμ 37 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Euh, 33, 334 était adopté Non, euh, c'était rejeté. Donc, donc amendement, 80, amendement 89. 89. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 90 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 335 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 336 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 91 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2 Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι τα 30 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 95 υπέρ. Όχι, όχι, λέει η πρόεδρος, έκανα λάθος, με συγχωρείτε. 94, 94 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 95 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 338 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 31 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. 96 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Amendement 339. Euh, 339 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Budget 38 38 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Φαμ 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άφε 32 υποπαράγραφος 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άφε 32 Ξεχωριστή ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τριάντα 39 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Άφετ 32 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 100 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Φαμ 40 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. ΦΑΜ 41 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. ΦΑΜ 42 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 342 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. ΦΑΜ 43 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 343 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 100 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Φαμ 40 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Αφε 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ΦΑΜ 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ΑΦΕ 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται άφε 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 344 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Αφετ 35 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Προϋπολογισμός 39 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 104 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Προϋπολογισμός 40 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Άφε 36 Ξεχωριστή ψηφοφορία, πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 105 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 348 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία υπαριθμών 7. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται να σηκώνετε τα χέρια σας ευκρινώς, αλλιώς δεν σας βλέπω. Οι άλλες καταπίπτουν. Προφορική 8, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Προϋπολογισμό 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 110 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολία 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άφετ 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 114 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. προφορική τροπολογία 6. Όχι. Όχι. Τροπολογία 116. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Budget 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 118 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ίντα 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ίντα 36. Άρχεται. Λείπει μία ψήφο. Λήξη τη πληροφορία. Εγκρίνεται. Τροπολία 119 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 352 έχει αποσυρθεί. Είναι τα 37 υπέρ. Είναι τα 37 υπέρ. Υπέρ λέω. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 120 Budget 45 πρώτα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 120. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 121. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 353. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 124 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. ΦΑΜ 45 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. ΦΑΜ 46 υπέρ. Κατά Αποχές απορρίπτεται. 125 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε καλά. Περνάμε στα παραρτήματα.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 Υιοθετείτε αυτόματα. Ωραία. 128 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Είναι τα 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρία 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι τα 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Είναι τα 40 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Συμβασμός 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Είναι τα 41 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται είναι τα 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Είναι τα 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμό 20. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Είναι τα 44 υπέρ. Κατά. Κατά, Εγκρίνεται. Τρακόσια υπέρ. Κατά Αποχές... Απολύπτωται. 371 υπέρ. Όχι, καταπίπτει. Αφέτ σαράντα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 372 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 373 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ...374... ...υπέρ... ...κατά... ...αποχές εγκρίνεται... Το ...τροπολογία 375 υπέρ... ...κατά... ...αποχές απορρίπτει... 135 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 376 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται είναι τα 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 377 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 3.78 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινε. 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 379 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 380 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 381 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 137 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 382 υπέρ. Κατά. εποχές Απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση 22. Χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά ε, εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 383 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 388 όχι καταπίπτει είναι τα 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 390 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Είναι τα 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 395. 393. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3.95 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Κατά πίπτη 399 αφέτ 43 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 141 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 142 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται Συμβασμός 25 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Είναι τα 53 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. Αφέτ 44 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. 401 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. τροπολία 145. Mm. Όχι. Κατόν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι τα 55 υπέρ. Κατά αποχές η ηλεκτρονική εξακρίβωση. Είναι τα 55. Άρχεται η ψηφορία. Λήξη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Φαμ 47 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός 26 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 402 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 56 κατά πίπτη, 405 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μετά 407 χωριστή ψηφοφορία η πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 408 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 147 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 148 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Είναι τα 57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται ηλεκτρονική εξακρίβωση. Για την ίντα 57. Ψηφίζουμε. Λήξη ψηφοφορία. Υιοθετήθηκε. Εγκρίνεται με μια ψηφοδιαφορά. Είναι τα 59. Υπέρ. κατά υιοθετήθηκε είπα ψηφίσαμε και την υιοθετήσαμε είναι τα 59 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται τροπολογία 149 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται είναι τα 60 Ψηφίσαμε την 58. Ε, σημείωσα ότι την υιοθετήσαμε. Αν θέλετε την ξαναψηφίζουμε. Ζητώ συγγνώμη. 58 ψηφίζουμε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελεκτρονική ηλεκτρονική ψηφοφορία. Le vote Λήξη πληροφορία. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. 59 την κάναμε, 149 την κάναμε. Είναι τα 60. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 409. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 410 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 151 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 411 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 412. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 153. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 154. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 155. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 413. Υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. ΦΑΜ 48 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. ΑΦΕΤ 46 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. ΑΦΕΤ 47 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 156 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 414 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 158 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 160 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 415 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 416 με συγχωρείτε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Είναι τα 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Φαμ 49 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 161 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Είναι τα 63 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ωραία, αν το θέλετε, είναι τα 63. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Με συγχωρείτε. Φαμ 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 162 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 163 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 417 υπέρ, κατά, αποχές, θέλω να ελέγξουμε, σας παρακαλώ. 417 υπέρ. Ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικά. 417 ελέγχουμε ηλεκτρονικά, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται με τρεις ψήφους. 418 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. ΦΑΜ 52 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Σαράντα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 164 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 419 υπέρ κατά αποχές Θέλω να ελέγξουμε ηλεκτρονικά σας παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε για την 419. Πέρας. Απορρίπτεται. 165 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 420 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 166 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 167 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 168 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι τα 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Είναι τα 64. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με τρεις ψήφους επιπλέον. Εκατόν εξήντα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εκατόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 421 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 171 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άφετ 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 172 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 422 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 173 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 174 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 175 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 423 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Alors, 60, 67 υπέρ, κατά, αποχές, δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα, άρα ελέγχουμε ηλεκτρονικά σας παρακαλώ, είναι τα 67, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Ανταπτή. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 27. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ίντα 68. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 180 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 427 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Φαν 54 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 428 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 182 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 193, 83 με συγχωρείτε υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 429 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 430 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Φαμ 53 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Φαν 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 434 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 435 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 29 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. «437 υπέρ» κατά «αποχές απορρίπτεται» Είναι τα 69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εκατόν ογδόντα έξι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. τα 70 υπέρ. Κατά. Εποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. τα 70. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται. Λείπει μία ψήφος. Πέρας. Εγκρίνεται. 187 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 443 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε βεβαίως ηλεκτρονικός έλεγχος επί της 443. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Φαμ 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 444 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβιβασμός 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 187 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προϋπολογισμός 48 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 188 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 33 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 455 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Προϋπολογισμός 51 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 188 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβασμός 34 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Προπολογισμός 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 456 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 457 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 459, πενήντα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προϋπολογισμός 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 460 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται προϋπολογισμός 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται προϋπολογισμή 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 35. Ξεχωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 461 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. προϋπολογισμοί 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 191. Ψηφίζουμε, λέει πρόεδρος, αναρωτιέται. Το Ι του 191 ψηφίζουμε μόνο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 465 υπέρ. Κατά κατά αποχές απορρίπτεται 191 το διπλό ή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προϋπολογισμή 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 466 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται φάν 58 πρέπει να την ψηφίσουμε. φάν 58 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. 468 και 192 468 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβασμός 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4, ε, συγγνώμη, συμβασμός 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 473 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 474 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 475 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 196 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 477 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται είναι τα 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 478 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται φαμ 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 198 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 199 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 200 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 479 υπέρ κατά α, αποχές απορρίπτεται 201 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 202 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 203 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 204 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άφετ 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 205 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 206 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 207 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 480 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 481 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται άφετ 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 208 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άφετ 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 209 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 200 84-85 Υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική εξακρίβωση. Άρχεται. Δύο ακόμα ψήφοι. Μία. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τέσσερα έχει αποσυρθεί. 213. Την ψηφίζουμε. 213 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άλλες 20 σελίδες έχουμε ακόμα. On fait un bloc, euh, d'accord. On fait amendement 214. Από το 2.14 στη 2.19 Τι ομαδοποιούμε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται όλες μαζί. 486. 487 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Να ψηφίσουμε την αιτιολογική σκέψη. Όχι. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Budget 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Budget 4. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Budget 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Φαμ 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Φαμ 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 22 αποσύρθηκε, είναι τα 1 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Φαμ 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Φαμ 5 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2.26 όχι, budget 6 και άφετε ένα μαζί. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται, απορρίπτονται. 2.26 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Αφετείο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Είναι τα δύο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. το 8. Υπέρ. Κατά εποχές απορρίπτεται άφετ 5 περ κατά εποχές απορρίπτεται τροπολογία 228 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται άφετ 4 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται συμβασμός 1 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Δύο υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία, προφορική τροπολογία 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Budget 9. Περ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Φαμ 6. Περ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6. Υπέρ Κάθε 6 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 2.35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Budget 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το ίδιο 35 απορρίφθηκε, άρα δεν καταπίπτει η budget 10. Ποιος είναι υπέρ της 10 κατά αποχές εγκρίνεται λοιπόν. Συμβασμός 2. Άφετε 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. ...2.39 απορρίπτεται... ...φάμε 7... ...υπέρ... ...κατά... απόχέ ...απορρίπτεται... Αφέτο 8... ...υπέρ... ...κατά... ...αποχές απορρίπτεται. Είναι τα τρία. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Μπάτζετ 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Είναι τα τέσσερα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται είναι τα πέντε. υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται φάμ 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβασμός 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ΦΑΜ 9 Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Αφέτ 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Φαμ 10. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Φαμ 11. Υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται φαμ 12 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται συμβασμός 4 υπέρ κατά εποχές Το πολίγιο 243 υπέρ κατά εποχές Απορρίπτεται. Είναι τα έξι. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Budget 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αφετέκα υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Φαμ 13 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Φαμ 14 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Συμβασμός 5 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Συμβασμός υπέρθμων 6. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 2.48. Όχι. Είναι τα 7 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Ε, εξακριβώνουμε ηλεκτρονική εξακρίβωση. Τροπολογία, τροπολογία 249. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απόχέ, απορρίπτεται. Συμβασμό 7 υπέρ, κατά, απόχέ, εγκρίνεται. Budget 11 υπέρ, ε, 15 συγγνώμη υπέρ, κατά, αποχέ, απορρίπτεται. Είναι τα 8 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Φαμ 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός υπαριθμών 8 τη ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Φαμ 16 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 18 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίθηκε. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Είναι τα 10. κατά Καταπίπτει. 2.55 έχει αποσυρθεί. Τροπολογία 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. ...2.56 έχει αποσυρθεί... Είναι τα 11. Μισό λεπτό. Η 38 της ΑΦΕΤ δεν έχει εγκριθεί. Ωραία. Τροπολογία 21 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 22. Υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε την έναρξη ε, δια, διοργανικών άτυπων διαπραγματεύσεων επί τη βάση των τροπολογιών που μόλις υιοθετήσαμε. Ποιο είναι υπέρ της έναρξης αυτών των διαπραγματεύσεων, κατά, αποχές. Να το κάνουμε ηλεκτρονικά. Λοιπόν, ψηφίζουμε για την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Έναρξη ψηφοφορία. Λοιπόν, είναι τέσσερις ψήφοι. Δύο τώρα. Λήξη ψηφοφορίας. 22 ψήφοι υπέρ, μία αποχή. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μπέρμαν για αυτό το τιτάνιο έργο. Ε, ε, Μάλιστα. Ε, προς ενημέρωσή σας, ορισμένοι από εσάς μπορεί να εξαπλάγησαν με το γεγονός ότι πολλές από τις τροπολογίες της Επιτροπής ΦΕΜ ε, απορρίφθησαν. Δεν είναι επειδή είμαστε αντίθετοι, αλλά δεν χρειάστηκε να τις ψηφίσουμε. Δεν υπήρχε λόγος να κρατήσουμε το νομοθετικό κείμενο ε, με όλες αυτές τις τροπολογίες. Έπρεπε να είμαστε σύντομοι, γι' αυτό τις απορρίψαμε. Λυπάμαι. Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ συγητή για τη δουλειά και θα ήθελα να του συστήσω να μην περιμένει μέχρι το τέλος των διαπραγματεύσεων για να μα αγοράσει τη σαμπάνια, να το κάνει ήδη απόψε. Πολύ καλή ιδέα. Φροντίστε το κύριε Μίτσελ, εσείς.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 αποχές εγκρίνεται. Προπολογία 31 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμό 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά αποχές νομίζω θα πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε επί της 33. Άρχεται η ψηφοφορία. Λείπουν τρεις ψήφοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ε, μπορούμε να πλαγάρουμε την 47. So το κάνουμε όσο το δυνατόν συχνότερα γίνεται. Μέχρι την 47, μπλοκ. Ψηφίζουμε από την 34 μέχρι την 47, συμπεριλαμβανωμένη στη 47, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 48 υπέρ, κατά Αποχές εγκρίνεται. 49. Ξεχωριστή και ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α, έχει απορριφθεί. Ας ελέγξουμε την 51. Έλεγχος. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται «55 και 56 μαζί ψηφίζουμε». Α, όχι, όχι, 55 υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 57 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τώρα ψηφίζουμε από κοινού από την 61 μέχρι την 63. Συμφωνείτε? Ωραία, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 64. Ξεχωριστή ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ. Ψηφίζουμε την 64. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 65 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Μπορούμε από κοινού να ψηφίσουμε από την 68 έως την 72. μέχρι την 72. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβιβασμός 4. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Από την 73 μέχρι την 75 όχι, όχι, την 74-75, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνονται. Συμβασμός 5, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Από κοινού, από την 77 μέχρι την 79, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνονται. Προφορική τροπολογία υπαριθμών 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ωραία, ελέγχουμε ηλεκτρονικά την προφορική υπαριθμών 2, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Με τέσσερις ψήφους διαφορά. 81 έως 83 έως 84. Μπερδεύτηκα τώρα, λέει η πρόεδρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 7. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Pardon, 88. 88 88 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 89. Ξεχωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 90 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 91, ξεχωριστή ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Μπορούμε να ψηφίσουμε από κοινού τις τρεις πρώτες της Επίτροπης Αλίας 1, 2 και 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Πες 4 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται πες πέντε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έξι επτά όχι όχι έξι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται επτά υπέρ ε, κατά αποχές Απορρίπτεται. Θέλετε έλεγχο. Με συγχωρείτε δεν ήμουν προσεκτική. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Αλία 7. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Όχι, θέλετε να ελέγξουμε. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πες 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πες 8. Ψηφίζουμε πέρας. Απορρίπτεται. με διαφορά δύο ψήφων. Δεν είναι σταθερές οι πλειοψηφίες. Πες εννέα. Πες εννέα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πες δέκα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πες έντεκα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πες 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πες 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πες 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πες 15 υπέρ Α, συγγνώμη, ξεχωριστή λέει. Α, έκανα λάθος λέει η πρόεδρος, δεν ξεχωριστή, με συγχωρείτε.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 ΠΕΣ 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 93 ξεχωριστή ψηφοφορία υπέρ του πρώτου κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 94 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 98 ξεχωριστή ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά αρχίζει η ψηφοφορία επί του δευτέρου τμήματος λείπουν δύο ψήφοι πέρας ισοψηφία, άρα απορρίπτεται. Alors, on, est, on fait vote bloqué. Ψηφίζουμε από κοινού. Είναι δύσκολο, είναι αρκετά δύσκολο. Όχι, όχι. 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε από κοινού την 104, από την 104 μέχρι την 108. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. «109. Ξεχωριστή πρώτο τμήμα υπέρ» κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 110 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 111 έχει αποσυρθεί 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβασμός 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 116 ξεχωριστή πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 117 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 118 και 19 από κοινού υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Προφορική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 121 έχει αποσυρθεί από 122 μέχρι 124 υπέρ. Όχι, δεν θέλετε. Καλά, καλά, καλά. 122-123 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 124 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 125 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 126. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 127 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Απασχόληση 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Απασχόληση 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Απασχόληση 3 ξεχωριστή πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Μπορούμε από κοινού να ψηφίσουμε μέχρι και την 9, αμπλουά 9, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 128. 128 με 132 από κοινού ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 133 ξεχωριστή ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ...134 έως 142 από κοινού υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Προφορική 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η προφορική φαμ 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Unblocked, από κοινού από φαμ 2 ψηφίζουμε μέχρι, μέχρι φαμ 20 μέχρι φαμ 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Προφορική 5 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Φαμ 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 με 26 από κοινού ψηφίζουμε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Στη συνέχεια, στην... από την 5 μέχρι τις 10 στις αιτιολογικές σκέψεις υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Προφορική 1 Προφορική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ωραία, αν θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο, ελέγχουμε την προφορική υπαριθμών 1. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. μπορούμε να ψηφίσουμε από κοινού από την 12 μέχρι τη 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 16 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε ηλεκτρονικά τροπολογία 16 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία 17 υπέρ Α, με συγχωρείτε 17 λέει η πρόεδρος μέχρι 27 αν συμφωνείτε όλοι από κοινού υπέρ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 Εντάξει, πέρας. Εγκρίνεται 21 ψήφοι υπέρ, 3 κατά και καθόλου αποχές. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία ε, Σνίμπερ Γιάστραμ. Κυρία Πρόεδρε, σύντομα, θα ήθελα να ευχαριστήσω εγκάρδια όλες τις επιτροπές που συμμετείχαν στη συζήτηση. Ε, θα ήθελα να το κάνουν αυτό και όλοι όσοι δεν συμμετείχαν και ελπίζω έτσι να είναι την επόμενη φορά. Τώρα τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κάρλος και τον συνεργάτη μου Μπάστιαν για την εξαιρετική και πολλή δουλειά τους. Ευχαριστώ. Alors, nous allons maintenant voter euh, sur le projet d'avis de Madame. Περνάμε στην ε, γνωμοδότηση της κυρίας Γκρέζ. Τροπολογία 1. Α, είναι ταυτόσιμες οι 1 και οι 2. Ποιος είναι υπέρ. Κα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Et nous votons donc euh, Ψηφίζουμε λοιπόν όλη τη γνώμη όπως τροποποιήθηκε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη ψηφοφορίας. 19 ψήφοι υπέρ, 5 κατά. Εγκρίνεται. Υιοθετείτε γνώμη. Yes. Um, on behalf of Mrs. Uh, Mrs. Εκ μέρους της κυρίας Κρέις ε, θα ήθελα να πω ότι θα ήθελε να γίνει γνωστό και να καταγραφεί στα πρακτικά ότι πλέον δεν υποστηρίζει αυτή την έκθεση. Sorry, for the avoidance. Ναι, προς αποφυγή αμφιβολιών. Δεν αποσύρει το όνομά τη από την έκθεση τη συγκατάθεσή της ΣΥΡΙ. Euh, Ωραία. Περνάμε στην ε, την μη νομοθετική γνωμοδότηση της ε, κυρίας Γκρές. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Όχι. Okay. ηλεκτρονική εξακρίβωση για την τροπολογία 1. Άρχεται ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Με δύο ψήφους διαφορά. Προφορική τροπολογία πίπτη. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά εποχές Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. εποχές Εγκρίνεται. Ηλεκτρονική εξακρίβωση. Τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Όχι. Η ψηφοφορία με πριν. Ωραία. Εξακρικοβώνουμε ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Με δύο ψήφους διαφορά. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται για 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε το σύνολο της γνώμης, νομοδότησης, ε, άρχεται η ψηφοφορία. Ένα άτομο δεν έχει ψηφίσει ακόμα. Λίγη ψηφοφορία. Ε, εγκρίνεται. 19 υπέρ, 5 κατά. Στην εισηγήτρια. Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ να καταγραφεί τα πρακτικά ότι η κυρία Γκρέζ δεν στηρίζει αυτή την έκθεση, ωστόσο θα θε, ήθελε να παραμείνει το όνομά της στην έκθεση καθ' αυτή. Έτσι για τελευταία φορά προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Μάλιστα, σημειώθηκε. Ça, c'est Mitchell. C'est la bonne euh, liste de vote. Euh. Oui, voilà, c'est ça. C'est le plus court, euh, le plus court d'aujourd'hui. D'accord. Voilà. Τώρα θα περάσουμε στην έκθεση Μίτσελ στην, για ε, τον προπολογισμό. Πρώτη προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. 3. Τροπολογία 3. Υπέρ. Να ελέγξουμε το νούμερο 2 γιατί μπερδευτήκαμε κάπως. Ευχαριστώ. Donc, on vérifie électroniquement l'amendement 2. Le vote est ouvert.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 Qui est contre Qui s'abstient Rejeté. Amendement 16. Qui est pour Qui est contre Qui s'abstient Rejeté. Amendement 5. Qui est pour Τροπολογία 5. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 6. Υπέρ, κατά, απόχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. από την 7 ως την 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, εγκρίνονται. Ε, Τιολογική σκέψη ο Όλα τα όλες οι τιολογικές σκέψεις μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Ψηφίζουμε στο σύνολο της νομοδότησης ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Ομόφωνα υπέρ. Μπράβο στην κυρία ε, Στρίφλερ. Τελειώσαμε τις ψηφοφορίες. Uh, ε, Jolie, can I... Κύριε Πρόεδρε, εκ μέρους της Επιτροπής θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας πλοηγήσατε ε, εν μέσω μιας πολύ δύσκολης ψηφοφορίας και το κάναμε και σχετικά σύντομα. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Τώρα, χωρίς να καμφθεί ο ζήλος μας, θα περάσουμε στην σημείο 20 της ημερήσιας διάταξης. Ανταλλαγή απόψεων για το σχέδιο έκθεση του κ. Νόιζερ Εργασίας Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ Ευρωπαϊκή Ένωση το 2011. Όπως γνωρίζετε είναι μια αιτήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης την οποία εκδίδουμε κάθε χρόνο και που ε, σχολιάζει τις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης το προηγούμενο έτος. Κύριε Νόιζερ, έχετε το λόγο για να μας παρουσιάσετε την έκθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σύντομος θα είμαι. Η ε, κοινή ΙΞΙΕ και ΕΟΥ συνεδρίασε στην Βουδαπέστη στην Ουγγαρία και το φθινόπωρο του 2011 στη Λαμέ του Τόγκο. Δέκα ψηφίσματα συνολικά ψηφίσαμε. Υπήρξαν διερευνητικές αποστολές στο Ανατολικό Τιμόρ, και στο Μπουζάν για την εξακρίβωση της ε, ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο Επίτροπος Πίμπαλξ είναι ο αρμόδιος επίτροπος και συμμετείχε και αυτός. Οι επιτροπές της ε, συνέλευσης ε, ΑΚΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεδρίασαν δύο φορές κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας της Βρυξέλλες και εδώ πρέπει να ασκήσω κριτική για την ε, χαμηλή συμμετοχή των Ευρωβουλευτών εδώ στις Βρυξέλλες. Η πλευρά της ΑΚΕ δικαίως ζήτησε οι επιτροπές να μην συνεδριάζουν πλέον κατά τη διάρκεια των τακτικών συνεδριάσεων του Ευρωκοινοβουλίου. Αυτή τη βδομάδα θα... Την Πέμπτη το μεσημέρι θα γίνει η πρώτη συνεδρίαση εκτός Ολομέλειας. Επίσης, κάπως ανησυχητική Σημαντικό ήταν ε, για την γραμματεία της ε, και Ευρωπαϊκής Ένωσης το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ορισμένα μέλη παρετήθηκαν τι θέσει τους και πρέπει να διασφαλιστεί η συνέχεια των εργασίων, μαλλή συνέχεια των εργασιών και Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προσπαθήσουμε ε, έτσι ώστε οι γνώσεις και οι εμπειρίε των συναδέλφων να μην χαθούν και να βρουν άξιους διαδόχους. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι το ζήτημα των βοηθών. Δυστυχώς υπάρχει μία επιφύλαξη στο ζήτημα των ε, βοηθών όσον αφορά την, ε, τις αποστολές της ε, συνελεύσεις και Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, η ομάδα εργασίας του 2011 ακολούθησε συγκεκριμένες μέθοδους εργασίας για τα ζητήματά της, καθορίστηκε ο πολιτικό ρόλο. αποφασίσαμε να ενισχύσουμε τον ε, πολιτικό μας ρόλο και την διαδικασία ε, αυτή. Υπήρξαν ορισμένες ε, τροποποιητικέ προτάσεις που διατυπώθηκαν το 2011 και ορισμένες από αυτές ψηφίστηκαν και πέρυσι, ορισμένες από αυτές μένει να ψηφιστούν φέτος. Θα ήθελα να τονίσω ότι η Συνέλευση και Ευρωπαϊκής Ένωσης θα γίνει ακόμα μεγαλύτερος, ε, ακόμα περισσότερο σημαντικός παίκτη στην περιοχή του Ειρηνικού και πρέπει να δώσουμε ειδικό πολιτικό βάρος στις θέσεις μας. Ταυτόχρονα, η ενασχόληση των, ε, της εξίε με ορισμένα πολύ σημαντικά ζητήματα χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια η κοινωνία των πολιτών ε, μεταξύ Βορρά και Νότου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μπορεί να κάνει τη διαφορά στην επίλυση τοπικών προβλημάτων. Επί τη ουσία θέλω να τονίσω ότι ο διάλογος ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Ευρωβουλευτές είναι ένα πάρα πολύ καλό όργανο το οποίο δεν θα οδηγήσει μόνο στην ε, δημιουργία κοινών θέσεων αλλά στην αλληλοκατανόηση και να σας ε, δώσω και ένα παράδειγμα με την Αραβική Άνοιξη. Το 2011 και στις δύο Ολομέλειες ασχοληθήκαμε με την Αραβική Άνοιξη εντονότατα και ε, αυτό είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει και στο μέλος. Επίσης, οι θέσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΑΚΕ είναι μέρη κοινέ και είναι σημαντικό να συνεχίσει ο διάλογος και σε επίσημο και σε ανεπίσημο επίπεδο. Και φυσικά είναι υψής της σημασίας να ε, χρησιμοποιούνται άκρως δημοκρατικές και διάφανες διαδικασίες κατά τη διάρκεια των ε, συνεδριάσεων, έτσι ώστε να λάμψει η δημοκρατική οδός ε, στην συνέλευση της και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, το 2011 ασχοληθήκαμε με ορισμένα πρόσθετα θέματα, με την μόλυνση των υδάτων, με την κατάσταση στην ακτή του ελέφαντος του, με το AIDS, με το χρέος με τους ανθρώπους με αναπηρία, την επιστημιστική κρίση στο κέρας της Αφρικής, ε, την κατάσταση ασφαλείας στην Σομαλία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ερυθρέα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Κύριε Κάσμαν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Νόιζερ για την εξαιρετικά καλή δουλειά που έκανε συντάσσοντας αυτήν την έκθεση. Θα ήθελα να θίξω δύο θέματα. Το ένα, το γενικό θέμα του διαλόγου. Με απασχολεί εδώ και αρκετό καιρό και με απασχολεί όλο ένα και περισσότερο αντί να είναι αντίθετο αυτό. Ιδιαίτερα η πλευρά της ΑΚΕ επιλέγει να μην ε, εισέρχεται σε διάλογο εάν δεν θέλει να συζητήσει και δεν, δεν της είναι ε, αρεστό το θέμα που προτείνουμε. Άρα δεν κάνει δούμε διάλογο. Γίνεται μονόλογος μόνο από πλευρά του. Και καταλαβαίνω ότι το ζήτημα της ε, μη διάκριση όσον αφορά την, ε, τις σεξουαλικές προτιμήσεις είναι ένα θέμα που ε, είναι πολύ άβολο για εκείνους. Εγώ εδώ σε αυτό το κοινοβούλιο έχω δει περιπτώσεις όπου παρότι το θέμα αυτό είναι στην ημερήσια διάταξη έχει προσπεραστεί με τους ρυθμούς και για να το ξεπεράσουμε, εγώ με τον Επίτροπο Πίμπαλξ οργανώσαμε μια κοινή ακρόαση. Σε αυτή την ακρόαση, η οποία είχε ως θέμα ε, το κοτονού ε, και την διάκριση με βάση τον κινητήσιο προσανατολισμό, πληροφορηθήκαμε από την ΑΚΕ ότι δεν θα συμμετείχε. Δεν υπήρχε εντολή για μη διάκριση βασισμένη στον γενετήσιο ε, προσανατολισμό για μένα σημαντικό είναι πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τον διάλογο, διότι εκείνοι μπορούν να φύγουν θέματα που τους ε, απασχολούν, όμως εμείς όχι. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει. Τώρα, το άλλο ευαίσθητο ζήτημα της ε, συνάντησης ΑΚΕ στο Σουρινάμ. Ο πρόεδρος αυτή τη στιγμή ε, βρίσκεται, ε, μάλλον για τον πρόεδρο εκκρεμούν πολλά εντάλματα συλλήψεως και ανάμεσα σε αυτά και ευρωπαϊκό εντάλμα σύλληψης. Και εγώ δεν θα πάω στο Σουρινάμ, αλλά η πρόθεση είναι όταν ο πρόεδρος ε, εκφωνήσει τον εναρκτήριο λόγο του, οι αντιπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποχωρήσουν. Όμως, εγώ πιστεύω ότι ο πρόεδρος θα χρησιμοποιήσει την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ε, υπονομεύσει αυτά τα εντάλματα σύλληψης, ιδιαίτερα το ευρωπαϊκό εντάλμα σύλληψης. Πιστεύω ότι είναι ανόητο, εξαιρετικά, διότι η εικόνα μας εδώ στην Ευρώπη θα αμαυρωθεί, θα θεωρηθούμε ασυνεπείς όσον αφορά τη στάση μας προς τον, την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Το είπα στον κύριο Νόιζερ, το συζητήσαμε και μου είπαν ότι η πλευρά της ΑΚΕ είπε ότι έτσι θα πράξουν, δεν θα αλλάξει τίποτα και λυπάμαι, αλλά για μένα ως Ευρωβουλευτή σε ένα κοινοβούλιο το οποίο έχει χτιστεί ε, στα θεμέλια της, ε, των ε, παγκόσμιων δικαιωμάτων και των ελευθεριών του ανθρώπου είναι απαράδεκτο να δεκτούμε μια τέτοια πρόταση. Ακόμα και σε αυτό το στάδιο λοιπόν θα ήθελα να, να παροτρύνω το Κοινοβούλιο να το ξανασκεφτεί. Το αναφέρω εδώ, ε, μη τηρώντας το πρωτόκολλο και παρακαλώ την ε, ανοχή σας, αλλά πραγματικά δεν θα μπορούσα να θίξω αυτό το θέμα στην ΑΚΕ χωρίς πρώτα να το έχω αναφέρει εδώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκέρενς έχει το λόγο. Ε, σε θέματα επιμελητίας καταρχήν, νομίζω ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε κατά πόσο μπορούν να παρευρεθούν και οι βοηθοί ή όχι, γιατί έχουμε σοβαρά έξοδα ταξιδιού και παραμονής. Γιατί ο βουλευτής θα αποφασίσει κατά πόσο χρειάζεται βοηθούς ή όχι, γιατί εκείνος καταβάλει τα έξοδα. Δεν είμαι ανήλικος, ίσως στο σπίτι μου, αλλά όχι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όσο αφορά την ουσία του προβλήματος, ο κύριος Νόιζερ είπε ότι οι χώρες ΑΚΕ είναι το σωστό φόρουμ για να ανταλλάξουμε αποφάσεις και να, λάβουμε, ε, να ανταλλάξουμε γνώμες, με συγχωρείτε, και να λάβουμε πολιτικές αποφάσεις με βάση τις συμφωνίες του Κοτονού. Γιατί έχουμε αρκετά στέρες βάσεις. Τώρα, το 2012, θα πρέπει να ξέρουμε κατά πόσο μπορούμε να διαιωνίσουμε αυτή την διάρθρωση, ναι ή όχι, των χωρών ΑΚΕ. Ενώ εγώ είμαι υπέρ της διάρθρωσης αυτής και όσο αφορά το Σουρινάμ, θα ήθελα να πω ότι εγώ δεν θα μεταβώ για τους ίδιους λόγους που προανέφερε ο Μάικλ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ζωζέ Κώστα Περέιρα έχει το λόγο εξ ονόματος της εξωτερικής υπηρεσίας. Επειδή είναι αργά και θέλω να περάσουμε σε μια άλλη έκθεση, του δίνω μόνο τρία λεπτά. Ναι, έχω συνηθίσει. Εμείς καλωσορίζουμε το σχέδιο ψηφίσματος γιατί πιστεύουμε ότι περιγράφει καλά τα αποτελέσματα των εργασιών για το 2011 και χρειάζεται πραγματικά να έχουμε και μια εξίσου καλή συνέχεια για αυτά που θεωρούμε τόσο σημαντικά ζητήματα. Όσον αφορά το σημείο 3 του σχέδιου ψηφίσματος, θα ήθελα να, ε, ε σας ε, τονίσω την προσοχή ότι το Συμβούλιο ότι όλα αυτά τα όργανα που αναφέρεται είναι ανεξάρτητα μεταξύ του, Συμβουλίο, Κοινοβούλιο κτλ. Ζητήθηκε να αντικατασταθεί η Προεδρία και η Προεδρία το δέχτηκε. Ως συνήθως, όμως, Η εσωτερική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωση έχει κάποιες συντηρήσει αυτό και αυτό με οδηγεί στο δεύτερο σημείο, το σημείο 3 του σχέδιου ψηφίσματο, το οποίο επιδοκιμάζει την επιστροφή του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη συμμετοχή στη συνέλευση ίσης εκπροσώπησης και μετά θα πρέπει να παρέμβουμε στις συνελεύσεις ίσης εκπροσώπησης όταν συντρέχει ο λόγος. Όλα αυτά σχετίζονται με το γεγονός ότι η ΕΙΑΔ είναι εκείνη η οποία θα πρέπει να θέσει εφαρμογή τον πολιτικό διάλογο, το άρθρο 96, τέτοιες περιπτώσεις και είμαστε από κοινού ε, υπεύθυνοι με την Κομισιόν όπως ορίζει, ορίζεται σε απόφαση του Συμβουλίου άρθρο 96 και μέσα στα πλαίσια της ε, ΕΙΕΔ. Σε σχέση με τους θα ήθελα να πω ότι στις 25 Ιουνίου 2012 ορίσαμε ένα νέο στρατηγικό σχέδιο ως προς τα δικαιώματα των γυναικών και του ρόλου τους και αναφερόμαστε στη συμμετοχή τους ιδιαίτερα σε μεταβατικές χώρες. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την ανασφάλεια και να προωθήσουμε την ανοικοδόμηση και να, πρέπει, και να προωθήσουμε και τη συμμετοχή και των δύο φίλων. Η ΕΙΕΔ μαζί με τα κράτη-μέλη και την Κομισιόν θα προσπαθήσουν να θέσουν αυτό το σχέδιο ενισχύ. Επίσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη στρατηγική εταιρική οικονομική σχέση μέσα στα πλαίσια ενός ολοένα και μεταλλασσόμενου κόσμου. Η συνέλευση ίσης εκπροσώπησης μπορεί να προωθήσει θέματα όπως την αηφόρο ανάπτυξη, κλιματικές αλλαγές, βιώσιμη ανάπτυξη και όλα αυτά θα τα κάνουμε μέσα στα πλαίσια αγαστής συνεργασίας και ζητώ συγγνώμη από τους διερμήνες γιατί μίλησα πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα, τόσο που δεν μπορούσαν να με παρακολουθήσουν. Ήταν αδύνατον. Ευχαριστούμε πολύ. Ο λόγος και πάλι στον κύριο Νόιζερ. Για δύο λεπτά μόνο. Εκτός μικροφώνου, κύριος Νόιζερ. Η ετήσια έκθεση του 2011 λοιπόν ήταν αυτή, ωστόσο θα ήθελα να τοποθετηθώ για το λεγόμενο πρόβλημα. Συζητήσαμε πάρα πολύ, σχεδόν ένα χρόνο για το θέμα του Σουρινάμ και της διεξαγωγής ε, της ε, συνελεύσης εκεί. Και στην Δανία, στο Χόλσενς, καταλήξαμε σε μια κοινή θέση. Και εμείς είμαστε οι διοργανωτές και εμείς θα αποφασίσουμε ποιος θα συμμετέχει και ποιος όχι στις ε, συνεδριάσεις μας. Έτσι λοιπόν δεν θα καλέσουμε τον πρόεδρο του, Σουριμάν, του Σουρινάμ, ωστόσο θα είναι παρόν. Και Παρότι εμείς ε, αποφασίσαμε και ε, όντως, όπως είπε και ο κ. Κάσμα, να εγκαταλείψουμε την αίθουσα αυτό, προσπαθήσαμε να του το μεταβιβάσουμε. Όντως είναι ένα πολύ προβληματικό ε, ζήτημα, όμως επειδή είμαστε κοινοβουλευτική συνέλευση ίσης εκπροσώπησης πρέπει να ακολουθήσουμε το τυπικό. Έχουμε κάνει παρόμοιες ενέργειες σε περίπτωση χωρών που δεν ακολουθούν δημοκρατικές διαδικασίες, όπως στη Ρουάντα για παράδειγμα ή στο, στην Κινσάσα του Κογκό. Ε, λυπάμαι κύριε Πρόεδρε, δεν μπορώ να αφήσω στο το τελευταίο σχόλιο. Αυτό που είναι μη δημοκρατικό για την ε, κυβέρνηση της Ρουάντα δηλαδή και το λέω ως κύριος παρατηρητής, ε, εκλογικός παρατηρητής των εκλογών του 2008. Πιστεύω πως είναι ακατάλληλο να προσπαθούμε να ε, δικαιολογήσουμε μία λάθος απόφαση και ο Νόρμπερτ, Νόρμπερτ δυστυχώς πρέπει να το το πω αυτό αλλά δεν είναι σωστό να κάνουμε συγκρίσεις με αυτές τις δύο χώρες, ιδιαίτερα συγκρίνοντας τη Ρουάντα και σίγουρα κανένα στη Ρουάντα, στην κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση δεν υπάρχει που να έχει ε, εκρεμές ένταλμα σύλληψης. Ευχαριστώ. Σας υπενθυμίζω ότι η προθεσμία ε, για τις τροπολογίες είναι 20 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι. Η ψηφοφορία θα γίνει στις 9 Οκτωβρίου. 12 λεπτά μένουν. Δεν αρκούν για να εξετάσουμε την επόμενη έκθεση. Κυρία Γκρές, κυρία υπέβαλε μια έκθεση που αφορά την ανάπτυξη των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε θέματα γενετικών πόρων και ιδιαίτερως τις επιπτώσεις τους στη μείωση της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες η διατηρήση, η διαχείριση και η ε, βιώσιμη ε, χρήση των γενετικών πόρων ε, καθώς επίσης και τα πλεονεκτήματα προσφέρουν αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε πρωτοσέλιδα. Θα, θυμηθεί, θα θυμάστε τα λευκά φασόλια της Βολιβίας για παράδειγμα. Αυτά τα θέματα συζητώνται από την κοινή γνώμη ιδιαίτερα η σχέση τους με τη γεωργία και την διατροφή, το, τη βιοειθική και το περιβάλλον, τη βιοτεχνολογία ε, και τα δικαιώματα του ανθρώπου. Λοιπόν, δίνω το λόγο στην κυρία Γκρέσ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους ε, συναδέλφους ε, που κατάφεραν να επιβιώσουν τις δυόμιση ώρες των ψηφοφοριών. Είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Θα ήθελα να σας πω ότι ως εισηγήτρια για αυτό το ε, θέμα πνευματικής διοκτησίας για τους γενετικούς πόρους και τις επιπτώσεις τους για τις αναπτυσσόμενες χώρες θέλω να, μα συγχαρώ όλους μαζί ε, όλα εμάς τα μέλη της ε, Επιτροπής ε, που, γιατί καταφέραμε να αναλάβουμε αυτή την το, πρωτοβουλίας το 90% της βιολογικής ανθρώπινης κληρονομιάς βρίσκεται σε ανεπτυσσόμενες χώρες, πλην όμως το 97% των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας τα κατέχουν επανεπτυγμένες βιομηχανικές χώρες. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μας ενδιαφέρει αυτό το θέμα και για ποιο λόγο ε, και το πώς οι αυτόχθονες ε, λαοί είναι στερημένοι και θύματα της βιοπειρατείας η έννοια αυτή ακούγεται λίγο ε, βάρβαρη, αλλά η πραγματικότητα είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστη, που κρύβεται πίσω από αυτήν. Πρόκειται για μια λαιλασία, βιομηχανική λαιλασία φυσικών πόρων και γνώσης ε, που βρίσκονται στις χώρες του Νότου. Πρόκειται για μια οικονομική και ηθική αδικία και μια απειλή εναντί της ε, βιοπικιλότητας. Μιλούμε για μια μάχη την οποία δίδουν οι ίδιες οι χώρες εδώ και αρκετά χρόνια. Γνωρίζω ότι δεν είναι η πρώτη φορά την οποία συζητούμε το θέμα αυτό εδώ. Θα θυμάστε την ανταλλαγή απόψε με την κυρία Άστον για το θέμα της βιοπειρατείας. Όμως είναι χρήσιμο να σας υπενθυμίσω ε, ενδεχομένως τον ορισμό ε, που μπορούμε να δούμε. Ε, είναι η ιδιωτικοποίηση και η εκμετάλλευση και η εμπορία, παράνομη εμπορία πόρων, βιολογικών πόρων ή παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται με αυτούς τους πόρους μέσω διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ε, από ιδιωτικές εταιρείε βιοτεχνολογίας και κυρίως χωρίς διαβούλευση ή αποζημίωση των λαών που ανέπτυξαν αρχικά αυτές τις γνώσεις. δεν μπορούμε να μιλήσουμε για βιοπειρατεία χωρίς να μιλήσουμε και για τους βιοπειρατές. Ποιοι είναι αυτοί οι πειρατές του ζών των οργανισμών που προερχόνται κυρίως από τρεις τομείς. Φάρμακοβιομηχανία, ε, καλλιντικά και αγροτροφημικό τομέα. Βγάζουν κέρδος στην πραγματικότητα από ε, πατροπαράδοτης γνώσεις ε, τις οποίες ε, τις ε, ονομάζουν, τις βαφτίζουν καινοτομία. Η εκμετάλλευση αυτών των γνώσεων δίνει σημαντικά κέρδη σε επιχείρησεις αυτές, ιδιαίτερα στον στη φαρμακοβιομηχανία, τα καλλιντικά και, την αγρο... και τον αγροτοφημικό τομέα. Ε, η... Τα προϊόντα των αυτόχθενων λαών ε, μάλλον αυτή η κατάσταση πραγματικά αποτελεί ε, μεγάλη μάχη και πρόβλημα για τους αυτοκτόνες λαούς. Η προστασία και η διατήρηση της ε, βιοπικιλότητας και της γενετικής ποικιλία ε, είναι κλειδί για τους στόχους χιλιετίας. Η γενετική πόρη είναι ιδιαίτερα σημαντική για μια βιώσιμη γεωργία και για την ασφάλεια των τροφίμων. Είπατε κι εσείς κυρία Πρόεδρε το παράδειγμα του λευκού φασολιού. Θα επανέλθω σε αυτό γιατί πραγματικά ε, ε είναι πολύ εύγλωτο. Ε, ο Λάρι Πρόκτορ, Αμερικανός πολίτης, ε, περπατάει σε μια αγορά στο Μεξικό μαζί με τη γυναίκα του, η οποία ονομάζεται Ινόλα. Ε, αγοράζει μερικά άσπρα φασό, ε, κίτρινα φασόλια, συγγνώμη, γυρίζει στις πολιτείες τα φυτεύει και το 1999 καταθέτει αίτημα για δίπλωμα ευρεσιτεχνία, το οποίο και παίρνει ε, για αυτά τα κίτρινα φασόλια του Μεξικού, που του δίνει το αποκλειστικό δικαίωμα ιδιοκτησίας αυτής της ποικιλία φασολιών. Είναι προφανές ότι ένας γεωργός του Μεξικού, ένας Μεξικάνος γεωργός, από εκείνη τη στιγμή και μετά ε, καταλήγει να πληρώνει δικαιώματα στον κύριο αυτό τον Αμερικανό για να καλλιεργεί τα φασόλια των προγόνων του. Αυτό το παράδειγμα, όπως σας είπα, είναι πραγματικά εύγλωτο ε, και ε, ε, κάνει πιο κατανοητό αυτό για το οποίο μιλάμε υπάρχουν δικαιώματα, διανοητικής ιδιοκτησίας επί των παραδοσιακών γενετικών πόρων ε, του ε, αναπτυσσόμενου κόσμου ε, που δημιουργούν πρόβλημα και στην και στην, που, που δημιουργούν δικαιώματα και στην, σε φάρμακα αλλά και προβλήματα στην πρόσβαση από πλευρά των αυξόμενου κόσμου. Ε, το θέμα αυτό είναι η βιοπειρατεία, δηλαδή είναι πρόβλημα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτές οι πρακτικές αντιβαίνουν ε, με τις ε, προθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκριζώσει την φτώχεια και να προστατέψει την βιοπικιλότητα. Επίσης αντιβαίνουν με την αρχή της λογικής συνέπειας της αναπτυξιακή πολιτικής ε, που αναφέρεται στο άρθρο 208 της Συνθήκης Λισαβόνα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά ε, είναι ταυτόχρονα ασυνεπές και το νομικό πλαίσιο διεθνώς. Ε, υπάρχει μια πολύ περίπλοκη αρχιτεκτονική με πολλά όργανα, διεθνή όργανα, ε, Οργανισμός Σωματικής Διοκτησίας, ο ΦΑΟ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου κλπ και χρειάζεται σίγουρα να ε, δουλέψουμε έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια συνολική και ενιαία ε, παγκόσμια διακυβέρνηση της χρήσης των ε, γενετικών πόρων. Πρέπει πρέπει να υποστηρίξουμε το σύστημα του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια και να βοηθήσουμε επίσης και τις αναπτυσσόμενε ε, χώρες που ε, εδώ και πολλά χρόνια προτείνουν πολύ απλά πράγματα. Τρία συγκεκριμένα. Πρώτον, ε, μια, ένα ρυθμιστικό πλαίσιο υποχρεωτικό που θα συνδέεται με τρία πράγματα. Πρώτον, να αναφέρεται η πηγή και η προέλευση των γενετικών πόρων και των παραδοσιακών γνώσεων που χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε εφεύρεση, σε εισαγωγικά εφεύρεση. Δεύτερον, να ε, αποδεικνύεται η ε, προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των αυτοχθών λαών και τρίτον, για τη χρήση των γενετικών του πόρων εννοώ, και τρίτον ζητούν την ε, δίκαιη και ισότιμη, το δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των κερδών. Είναι πολύ σημαντικό για μας εδώ σε Επιτροπή να γίνουμε αντιπρόσωποι αυτών των χωρών εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να γίνουμε η φωνή τους. Το μήνυμα είναι σαφές. Πρέπει η Σύμβαση Βιοπικιλότητας και το πρωτόκολλο της ε, Ναγκόγια να μπουν στο επίκεντρο της δράσης ε, και όλα τα υπόλοιπα να εξαρτηθούν από αυτή τη σύμβαση. Γιατί αυτή η σύμβαση επιτρέπει να εξασφαλίσουμε μια ισορροπία ανάμεσα σε ανεπτυγμένες και ανεπτυσσόμενες χώρες ως ε, Επιτροπή Ανάπτυξης θα πρέπει να συνεχίσουμε να ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη της ε, να επικυρώσουν γρήγορα το πρωτόκολλο της Ναγκόγια προκειμένου να καταπολεμήσουμε τη βιοπειρατεία και να ανακτήσουμε την δικαιοσύνη στις ανταλλαγές των γενετικών πόρων. Τέλος, η βιοπειρατεία ε, έχει τις ρίζες της στην ανεπάρκεια ε, νομοθεσία στι ίδιε αναπτυσσόμενε χώρε και στην απουσία μηχανισμών ελέγχου στις αναπτυγμένες χώρες. Μην ξεχνάμε επίσης και τον θεμελιώδη ρόλο που παίζει η αναπτυξιακή συνεργασία, η αναπτυξιακή συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που προτείνει που θα μπορούσε να προτείνει στις αναπτυσσόμενες χώρες βοήθεια για την ενίσχυση των μηχανισμών τους ε, που θα βοηθούσαν στην ειδική κατανομή των ε, κερδών, των ωφελών. Ε, είμαι ανοιχτή σε συζήτηση με, τις, με τους συναδέλφους των άλλων πολιτικών ομάδων έτσι ώστε πραγματικά να αποτελέσουμε ε, ε, να γίνουμε κήρυκες ε, της γνώμης των εψόμενων χωρών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε λίγα λεπτά. Ο κύριος Νόισερ έχει δύο λεπτά, το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ ως και ο να σας συγχαρώ για την πραγματικά καλή έκθεση. Εμείς ως ε, ομάδα των σοσιαλιτών στον θα ακολουθήσουμε μια ξεκάθαρη πολιτική γραμμή. Δύο πράγματα αναφέρονται ξέχω, ε, τη βιοπειρατεία. Είναι τα ένα από αυτά. Και σε γενικέ γραμμές υποστηρίζουμε πλήρως την εκθεσή σας. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν έχει το λόγο. Η κυρία Μπάρμπαρα Νόρκρος έχει το λόγο. <clears throat> Τρία λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω πως καλύτερα να συνεχίσω στα αγγλικά. Θα είμαι σύντομη. Βλέπω το χρονόμετρο και πέφτει. Λοιπόν, πιστεύω πως εμείς και από τη Γενική Διευθύνση Trade και από το DG Trade για ζητήματα εσωτερικής αγοράς, αν και λείπουν, νομίζω πως μπορώ να μιλήσω και εξ ονόματός τους, θα λάβουμε σοβαρά υπόψη όλα αυτά που έγραψε η κυρία Γκρέζ. Υπάρχει πολλή αλήθεια σε αυτά που λέει. Από την άλλη όμως μπορώ να πω ότι η Επιτροπή κάνει τη δουλειά της, μελετά, διαβάζει. Και οι συνάδελφοί μου στο GG περιβάλλοντος έχουν δεχτεί μία ε, εκτίμηση αντικτύπου για την κατάσταση και ελπίζουμε ότι στις αρχές Οκτώβρη θα υιοθετηθεί η νομοθετική πρόταση και μετά θα μεταφερθεί και στο, θα μεταβιβαστεί στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο πολύ γρήγορα. Φυσικά η κύρωση του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια επιφέρει και εφαρμοστικά και εκτελεστικά μέτρα που θα επιτρέπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να το υπογράψει και να το επικυρώσει. Αυτά τα μέτρα θα προετοιμαστούν πολύ γρήγορα, πιστεύω, και Ελπίζουμε την ίδια μερομηνία να έχουμε και την υιοθέτηση αυτών των μέτρων. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρουμε, όμως στο προσεχές μέλλον, στο πολύ προσεχές μέλλον θα γίνει αυτό. Έτσι λοιπόν το χρονοδιάγραμμα είναι λίγο πολύ αυτό. Ελπίζω πολύ γρήγορα να μπορέσουμε να επικυρώσουμε και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους για τη δουλειά τους. Εσείς ως Κοινοβούλιο έχετε τη δυνατότητα να συζητήσετε διεξοδικά το κείμενο νομοθετική, τη νομοθετική πρόταση και είμαι σίγουρη ότι όλοι μαζί και μαζί με το Συμβούλιο θα μπορέσουμε να βρούμε κάτι ουσιώδες. Το πρωτόκολλο είναι πάρα πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα σε αυτά που ζητάτε εσείς και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως έτσι κι αλλιώς πράττει τα τελευταία χρόνια σε όλες τις συζητήσεις σε διεθνές, διεθνή κλίμακα. Είναι ενεργικά συμμέτοχος και κάνει ό,τι μπορεί. Και το λέω αυτό γιατί σε πολλούς από αυτούς τους διεθνείς οργανισμούς χρειάζεται συνένεση, ιδιαίτερα στο θέμα του γενετικού, των γενετικών πόρων. Κάναμε μια πρόταση το 2005 σχετική, αλλά επειδή υπάρχουν αυτές οι διαφορετικές απόψεις, είμαστε κάπου στη μέση και αυτή τη στιγμή κολλιόμεθα κάπως. Γίνονται προσπάθειες νομίζω αυτή την εποχή για να ξεπεράσουμε αυτή τη διχοτόμηση και νομίζω το Δεκέμβριο θα προσπαθήσουμε να δούμε αν μπορούμε να καταλήξουμε σε έναρξη διαπραγματεύσεων από το 2013 και μετά. Θέλουμε να είναι το θέμα αυτό, να παραμείνει στην ημερήσια διάταξη, θέλουμε να σας υποστηρίξουμε. Όμω, όπω σα είπα, ε, πολλοί είναι οι διεθνεί οργανισμοί που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Σα υπενθυμίζω ότι στις 6 Δεκεμβρίου ε, θα εγκριθεί η έκθεση και στις 18 Οκτωβρίου μέχρι τις 6 το απόγευμα πρέπει να έχουν υποβληθεί τροπολογίες. Λυπάμαι ιδιαίτερα, αλλά επειδή έχουμε υπερβεί το χρόνο μας, δεν θα μπορέσουμε να δούμε το τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης, που ήταν η έκθεση του κυρίου Σβένσον, για την ε, στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να γίνει ανταλλαγή απόψεων πριν από την ψηφοφορία κατά την προσεχή μας συνεδρίαση και σας υπενθυμίζω ότι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι 5η 20 Σεπτεμβρίου στις 12 ε, το μεσημέρι για την έκθεση Σβένσον. Θα ξαναβρεθούμε εδώ στις 8 Οκτωβρίου από τις 3 μέχρι τις 6.30 και στις 9 Οκτωβρίου από τις 9 μέχρι τις 12.30 και από τις 3 μέχρι τις 6.30 το απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας και για την υπομονή σας. Καλό βράδυ.